η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο καταλόγους χωρών και οι δύο απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πρωτοβουλία μεταξύ άλλων της δικιάς μου πολιτικής ομάδας γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτοί που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τώρα να συμπεριλάβει και τον Παναμά και τη Σαουδική Αραβία. Αλλά για άλλη μια φορά, για να αναλύσουμε τον κατάλογο, θα έπρεπε να προσέξουμε ποιες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται. Αυτές κυρίως που δεν συμπεριλαμβάνονται, που δεν αναφέρονται στον κατάλογο. Τι γίνεται με την Ελβετία η οποία παραβιάζει κατάφορα διάφορα άρθρα του κώδικα της ομάδας που ασχολείται με την καταπολέμηση εισόδων από νομοποίηση εισόδων από Οπότε το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, πώς θα σταματήσει. Για να σταματήσει πρέπει να σταματήσουν και η φορολογική παράδειση, εκεί όπου κρύβονται οι μεγάλες περιουσίες των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα δημοσιεύσει ένα μαύρο κατάλογο, μια λίστα για χώρες που κάνουν ανακύκλωση ανεπαράλογο ναι, διότι ε, δεν ακολουθήθηκε μια αυτόνομη και ανεξάρτητη διαδικασία για να εξολογηθούν οι χώρες αυτές που ε, είναι απειλές όσον αφορά την εγκληματικότητα. Μετά από διάφορες απορρίψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά δημιούργησε έναν κατάλογο ε, που δεν είναι εξαντλητικό, με μεθοδολογία που είναι κάπω ή ανεξάρτητη. Η δημοσίευση τη νέα μαύρη λίστα είναι ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να θεωρηθεί μόνο σαν ένα πρώτο βήμα. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρε αυτού του καταλόγου είναι υπόκεινται σε πιο αυστηρού ελέγχου τη στιγμή που ασκούν δραστηριότητε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπάρχουν στρατηγικέ ελλείψει όσον αφορά την καταπολέμηση τη ανακύκλωση χρήματο και τη χρηματοδότηση ε, των τρομοκρατών. Πρέπει να γίνουν πολλά να εξασφαλίσουμε ότι όσοι δραστηριότητε πιέσεω που ασκούνται από τα λόμπι σε κάποιε χώρε να μην εξωτερώνουν τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να δρουν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Τέλος, είναι απαραίτητο η διαδικασία να γίνει ακόμα πιο διαφανής. Γι' αυτό ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διπλασιάσει τις αξιολογήσεις όσον αφορά τις χώρες που είναι στον κατάλογο για να υπάρχει και δημόσιος έλεγχος. Χαίρομαι ότι διότι πριν ολοκληρωθεί αυτή η θητεία έγινε άλλο σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την καταπολέμηση της ανακύκλωσης του χρήματος. Είναι φρικτό έγκλημα που εμπλουτίζει τους εγκληματίες ε, και που δρούν παράνομα. Είναι ένα έγκλημα που θα πρέπει να κατασταλεί και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατά διάκριση όπως και η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος επιτρέπει ποινικέ ε, ποινές και να είναι πιο αποτελεσματική δίωξη αυτών των εγκλημάτων. Δάτω μας για να καλέσω τα κράτη-μέλη εκ νέου να κάνουμε ταχεία και σωστή εφαρμογή του κειμένου στις εθνικές ενόμες τάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Ράντεφ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριε και κύριοι, το άρθρο 9 της 4ης και της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της χρηματοδότησης της δημοκρατίας ζητά από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν να διεξαγάγει ανάλυση του θεσμικού και νομικού πλαισίου των ε, χωρών εκτός Ένεσης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των, συστό, των συστημάτων τους ώστε να εντοπίζονται και να προσδιορίζονται ελλείψεις για τους στόχους αυτού της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλήματος χρήματος. Αυτά όλα είχαν συμφωνηθεί από όλα τα θεσμικά όργανα και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κανένα κράτος μέλος δεν είχε εκφράσει αντίρρηση. Να είμαι σαφής, η Κομισιόν είχε δημοσιεύσει χώρες υψηλού κινδύνου και στο παρελθόν που ήταν ε, ταυτόσιμες με εκείνες που περιλαμβάνονταν στους αντίστοιχους καταλόγους της Task Force. Αυτή τη στιγμή πλέον η Κομισιόν έχει ε, υποχρέωση να διεξαγάγει τη δική της αυτόνομη οικονομική ανάλυση που θα είναι ξεχωριστή από εκείνη της Task Force. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τεράστια ενιαία αγορά και πρέπει η Κομισιόν να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσει για όλε τις απειλές και αυτές που απορρέουν από ε, εξωτερικούς παράγοντες και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχο ε, κεφαλαιοκών ροών από έξω προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κεφαλαιακές ροές είναι ύποπτες ή ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι επιχειρηματικέ δραστηριότητες και συναλλαγές με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Απλώς αποτελεί ένα ε, προειδοποιητικό σημάδι να υπάρχει επαγρύπνηση διότι αν... Συγγνώμη, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω και εγώ να συγχαρώ τους συναδέλφους για όλη τη δουλειά που έχουν ε, κάνει οι κομισιόν, οι υπηρεσίες κομισιόν για τον προσδιορισμό χωρών ε, ε, υψηλού κινδύνου. Ξέρουμε πολύ, πολύ καλά όλοι μας πόσο σημαντικά είναι αυτά τα προβλήματα για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι χώρες που λειτουργούν ως φορολογική παραδιστή, είδου είδους κινδύνους δημιουργούν οι χώρες αυτές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό συμμερίζομαι όλες τις επιδιώξεις και αυτά που είπε η Επίτροπος είναι κάπως περίεργο. Είμαστε μια ένωση που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, στο κράτος δικαίου και ταυτόχρονα βλέπουμε το Συμβούλιο, ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα, να υποσκάπτει αυτή την, την αρχή. Δηλαδή την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία έχουμε συναποφασίσει. Θεωρώ ότι είναι μια καταστροφή, ότι είναι ένα σκάνδαλο πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που βλέπω ε, στο Συμβούλιο είναι ε, υπάρχει ένα μαύρο κουτί. Δεν ξέρουμε τι λέει το κάθε κράτος μέλος της ομάδας εργασίας και στις συνεδριάσεις αυτών. Πρέπει να απαιτήσουμε από το Συμβούλιο να γίνει καθαρό, να γίνει διαφανές, ώστε να μπορούν ε, και εμείς και τα μέσα ενημέρωσης να γνωρίζουμε ποιος, ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι που οδηγούν στο μπλοκάρισμα αυτής τη λίστα, τη μαύρης λίστας. Διότι αν δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίε, δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε μια αποτελεσματική και αποδοτική λύση και δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή την τόσο σημαντική του κράτους δικαίου που όλοι υποστηρίζουμε. Το λόγο έχει ένα λεπτό ο Σίρντεβαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να εμπλουτίσω τη συζήτηση αυτή με ένα πρακτικό παράδειγμα. Κάθε χρόνο, το έχουν αποδείξει αυτό ε, πολλές μελέτες, ε, εισραίουν ε, εγκληματικά κεφάλαια στον κατασκευαστικό κλάδο της Γερμανίας. Αυτό έχει ως ε, ε, πρώτο αποτέλεσμα βεβαίως να αυξάνει τις τιμές των ακινήτων και τα ενίκια κατά συνέπεια. Αυτό με τη σειρά του έχει την, το αποτέλεσμα ε, εκείνοι που πλήττονται από την πολιτική αδράνεια του Συμβουλίου να είναι οι ενοικιαστές, οι απλοί πολίτες. Και αυτός θα ήταν και από μόνος του λόγος να θεωρηθεί σκάνδαλο η απόρριψη της ε, λίστας από, την, ε, από το Συμβούλιο. Μπορεί κανείς να πει ότι το έργο της Κομισιόν δεν ήταν επαρκές, αλλά πάντως ήταν κάτι, μια αφετηρία πάνω στην οποία μπορούσαμε να βασιστούμε. Αυτό το μήνυμα πρέπει επιτέλους να το λάβουν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Thank you, Mr. Chair. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Η καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο, του εργανομένου εγκλήματο, τη φορολογική απάτη, απάτης είναι βασική προτεραιότητα όλων των πολιτισμένων χωρών στον 21ο αιώνιο αν και ίσω ο κύριο Κόμπαν μπορεί να διαφωνήσει. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολιτισμένε χώρε. και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει αυτά να αποτελέσουν προτεραιότητά μα. Αλλά ταυτόχρονα λέω ότι θα ήθελα να είναι προτεραιότητά μα. Δυστυχώ έχουμε μεγάλη απογοήτευση σήμερα. Η μεγαλύτερη απογοήτευση που, έχω, που είχα εδώ και αρκετό καιρό και δεν είναι λίγο αυτό που λέω. Η πλειοψηφία των κρατών μελών στο Συμβούλιο απέρριψε την μεθοδολογία ε, που, που, την, τη λίστα μάλλον που βασίστηκε πάνω σε στοιχεία και σε πολύ ορθή μεθοδολογία. Φυσικά η λίστα αυτή δεν ήταν τέλεια αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αφετηρία μια καλή διαδικασία στην οποία θα μπορούσαμε και εμεί να εκφράσουμε την άποψή μα σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το αποτέλεσμα και θέτει ένα αμφιβόλο την αφοσίωσή μα, την προσήλωσή μα, τι αρχέ μα και την αυτοπεποίθησή μα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να συνεχίσει το έργο τη και να ζητήσω από το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του και να σταματήσει να μα ντροπιάζει. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μορέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια μαύρη λίστα για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και τι μαθαίνουμε σήμερα, και το μαθαίνουμε με φοβερή απογοήτευση, ότι το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο ξεκάνει αυτό τον κατάλογο που δεν θέλει να βάλει στον κατάλογο αυτό χώρες οι οποίες είναι πασίγνωστο ότι είναι πρωταθλήτριες σε αυτού του τομεί. Παράδειγμα, πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί σήμερα ότι χώρες όπως ο Παναμά, η Σαουδική Αραβία συμμετέχουν σε αυτό το φαινόμενο με πραγματικά κλιματικέ πράξεις, όταν οι Ευρωπαίοι ζητούν περισσότερη ε, διαφάνεια. Μα με τον Παναμά ξέρετε τι η διερεύνηση έγινε και πώ καταλήξαμε στο ότι όντω υπήρχε ξέπλυμα και για τη Σαουδική Αραβία, είναι πασίγνωστο ότι οι ιδιώτε χρηματοδότησαν την Daesh, το ISIS. Οπότε τη διαπιστώνουμε αποτυχία. Το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο καταστρέφει την προσπάθεια αυτή. Εμείς πρέπει να καταγγείλουμε ως Κοινοβούλιο αυτή την κατάσταση. Μέρα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, το Συμβούλιο απορρίπτει τον κατάλογο. Κακός. Πώς θα εμποδίσουμε την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Κάτι το οποίο πρέπει να είναι στρατηγική για μας. Γι' αυτό και είχαμε και την οδηγία για την καταπολέμηση νομοποίησης παρανομού χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μπορεί να εντοπίσει τρίτες χώρες που βρίσκονται σε τέτοιο κίνδυνο και να εντοπίσει τις ε, αδυναμίες τους. Ο κατάλογος μπορεί να μην είναι τέλειος, είναι όμως αναγκαίος. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι. Πρέπει βέβαια στις χώρες που περιλαμβάνονται να δοθεί και ο χρόνος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση των συστημάτων τους και να μην συμπεριλάβουμε ε, τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ με τις μεταρρυθμίσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρακολουθεί τις 23 χώρες και άλλες και να χρησιμοποιεί τα μέσα που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι μονάδες της να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και όταν υπάρχει κάποια αλλαγή να μπορούν να προσαρμόζουν τον κατάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει κατάλληλους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει ε, και να υποστηρίξει και τα συμφέροντα τρίτων χωρών που δεν θέλουν να συνδεθούν με το φαινόμενο της νομοποίησης παράνομου χρήματος εφόσον όντω το αξίζουν. Και έπειτα υπάρχει το θέμα της Ρωσίας. Η Λίμπε, η Έκον και η Τάξη 3 ξανά και ξανά έχουν πει ότι η Ρωσία δεν προσαρμοζεται, δεν συμμορφώνεται με το οικονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει η υπόψη της αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το λόγο έχει ο κύριος Φαρία για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα δημοσιονομικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προστατεύονται και να μην επιτρέπεται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν τέτοιο κατάλογο που να βασίζεται βέβαια στην ανάλυση κινδύνου. Όταν υπάρχουν υποψίες πρέπει να ε, διαρευνώνται. Πρέπει να παρακολουθούμε τις συναλλαγές και σύμφωνα με την Europol μπορέσαμε να έχουμε μικρότερη απειλή, να έχουμε αναλύσει τις ύποπτες περιπτώσεις. Τώρα, δεν υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις. Καθ' άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνείται τον κατάλογο αυτό χωρών το Συμβούλιο. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε την νομοποίηση εισόδων από παράνομη δραστηριότητα. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένο βέβαια από αυτήν την ενωσιακή μαύρη λίστα. Αλλά παρόλα αυτά τα επιχειρήματά μας δεν θα πρέπει να οδηγούν στον αποκλεισμό χωρών που ξέρουμε ότι προχωρούν σε τέτοιες πρακτικές. Πρέπει να καταπολεμηθεί λοιπόν η νομοποίηση παράνομου χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εμείς θέλουμε να κλείσουμε τα κενά με κοινή λογική. Καλύτερα να προλαβαίνουμε. Προχωρούμε στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Έχω δεχθεί τρία αιτήματα. Γίνονται και τα τρία αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, η νομοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή πρέπει να χτυπηθούν. και αφού πίστηκε η επιτροπή επιτέλους να διαμορφώσει τη μαύρη λίστα των χωρών που φοροδιαφεύγουν βλέπουμε ότι το συμβούλιο αρνείται να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία μπλοκάρει πραγματικά την έκδοση της μαύρης λίστας των χωρών της φοροδιαφυγής. γιατί; επειδή εκεί είναι ο παναμάς; επειδή είναι η σαουδική αραβία. από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα διαφάνειας. όταν λέμε το συμβούλιο ποιες χώρες εννοούμε; όλες οι χώρες στο συμβούλιο ήταν αυτές που αρνήθηκαν να επικυρώσουν τον κατάλογο της κομισιόν; αν όχι θέλω να μας πείτε ποιες ήταν οι συγκεκριμένες χώρες οι οποίες έφεραν τα εμπόδια διότι πίσω από τη λέξη συμβούλιο υπάρχει μια πλήρης αδιαφάνεια και καλύπτονται συγκεκριμένες χώρες και πολιτικές. θέλουμε μια απάντηση κυρία κοτ στο θέμα αυτό πολύ συγκεκριμένη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μπιλμπάου Μπαράντικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στον κατάλογο αυτό δεν υπάρχουν όλοι, αλλά υπάρχουν αρκετοί. Συγχαρητήρια στην Επίτροπο και στην Επιτροπή. Έχει τη δικιά μας στήριξη. Η στάση του Συμβουλίου είναι ατυχέστατη. Και γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μας. Και δεύτερον, γιατί μας ζημιώνει όλους. Ό,τι είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καλό για όλες τις χώρες μέλη και δεν υπάρχει διαφάνεια. Το επαναλαμβάνουμε, οι χώρες μέλη κάνουν παζάρια μεταξύ τους για να προστατεύσουν τα δικά τους μεμονωμένα συμφέροντα, τα βρίσκουν μεταξύ τους και τελικά δεν υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τη συλλογική θική. Πρόκειται για πρακτικές οι οποίες ζημιώνουν τους πόρους που διαθέτουμε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τελικά είναι οι χώρες μέλη που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνει με το κύρος της. Μα έτσι τρέφεται ο λαϊκισμός. Οπότε γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την εκπρόσωπο του Συμβουλίου για ποιους λόγους απορρίψατε τον κατάλογο. Πείτε μας, αν μη τι άλλο, δύο λόγους. Το λόγο έχει ο κύριος Θέριτς για ένα λεπτό. You didn't ask the floor. You have the floor. Δεν ζητήσατε το λόγο. Τον έχετε. Παρακαλώ. Sorry, Mr. President, Συγγνώμη, ε, δεν κατάλαβα τι είπατε. Εξαιρετική ιδέα. Καταπολέμηση τρομοκρατία. Κανεί, μα κανεί δεν είναι περισσότερο υπέρ τη καταπολέμηση τρομοκρατία από μένα. Απολύτω. Πρέπει επιτέλου να ξεκινήσουμε. Πρέπει επιτέλου να του σταματήσουμε ε, το, το ξέπλυμα χρήματο στη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Όλα αυτά. Αλλά περιμένετε. Συνειδητοποιώ ότι η όλη συζήτηση πολλές φορές επαναφέρει στο, ότι, στο το γεγονός ότι δεν, δεν μπορείς να υπησέλθεις σε πολύ μεγάλο βάθος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο τραπεζικό σύστημα και μετά είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, να, να τα ρίχνεις όλα ε, στους κακούς, στη Ρωσία κτλ. Βεβαίως, Μήπω όμω χρειάζεται περισσότερο ε, οι τραπεζικέ αρχέ, οι χρηματοπιστωτικέ αρχέ να έχουν περισσότερε αρμοδιότητε για να ελέγχουν τραπεζικού λογαριασμού. Είμαι λίγο καχύποπτο λοιπόν. Καταπολέμηση τρομοκρατία, ναι, είναι θετικός ε, στόχος, αλλά νομίζω ότι ε, κρύβονται λίγο περισσότερα πράγματα. Μήπω θέλετε να βλέπετε τους ε, τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο όνομα τη Επιτροπής, το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ που με το λόγο, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Αυτή είναι η πρώτη φορά πράγματι που επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατάλογο που περιέχει χώρες υψηλού κινδύνου. Και όταν συζητήσαμε τη μεθοδολογία και σχεδιάζαμε την προσέγγιση και τη λογική και τα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση. Το ξέραμε τότε ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, θα ήταν κάτι απαιτητικό. Από πλευρά τεχνογνωσία θα ήταν ευαίσθητο θέμα, διότι εργαζόμαστε στο πλαίσιο γεωπολιτικών και εξωτερικών δεσμών και επαφών που έχει κάθε κράτος μέλος. Ε, ξέραμε ότι ίσως δεν θα ήταν κάτι δημοφιλές, αλλά ξέραμε σίγουρα, πραγματικά, ξέραμε ότι είναι κάτι αναγκαίο, διότι αυτές οι χώρες, οι τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου είναι ένα σημαντικό στοιχείο ε, σχετικά με ό,τι κάνουμε κατά του ξεπλήματος χρήματο και της χρηματοδότησης των τρομοκρατών, είναι ένα σημαντικό στοιχείο όλου του συστήματος και θα το επαναλάβω εκ νέου ότι αυτό κάνουμε στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι όσον αφορά τη συστηματική πρόληψη. Αυτό αφορά πρόληψη αυτό που κάνουμε. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του πώς είναι διασυνδεδεμένος ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Αν θέλουμε να έχουμε έναν ασφαλή οικονομικό τομέα, δεν πρέπει να αφήνουμε ασθενή σημεία και εύκολα σημεία εισόδου στο σύστημα εκ των έξω. Όποτε συζητώ αυτά τα θέματα με τις αρχές επιβολής του νόμου, με τους εμπειρογνώμονες και εκείνους που εφαρμόζουν όλα αυτά τα συστήματα, πάντα έχουν σαφέστατο στόχο που μας θέλουν κόψτε την εισρωή παρανόμου χρήματος στην Ευρώπη, διότι αυτό είναι το χρήμα το οποίο ε, χρηματοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και την ε, τρομοκρατία. Αυτό κάνουμε λοιπόν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι χώρες που έχουμε στον κατάλογο ανήκουν στον κατάλογο. Ταυτόχρονα ε, βλέπουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα, διότι ήταν στο επίκεντρο των επικρίσεων που ακούσαμε από τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ. Ίσως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Το άκουσα αυτό να αναφέρεται και εδώ στο Κοινοβούλιο στη σημερινή συζήτηση ότι θα θέλατε να δείτε λεπτομερέστερη αξιολόγηση. Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια και χρειαζόμαστε ισχυρό καλύτερη υιοθεσία, αν θέλετε, να τα εστερνιστούν τα κράτη-μέλη πλήρω. Θα πρέπει να ελέγξουμε εκ νέου κατά πόσο τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να συνεργαστούν και κατά πόσο ε, τελικά υπάρχει, ε, ε, δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον την καταπολέμηση των και των οργανωμένου εγκλήματο από τα κράτη-μέλη. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα δούμε ότι υπάρχει ετοιμότητα από πλευρά κρατών μελών διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο σύστημα αυτό όπου τα οικονομικά ιδρύματα και το χρηματοδοτικό σύστημα αυτό ε, δεν έχει σύνορα. Δεν έχει σύνορα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτο μέλο δεν μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο. Πρέπει αυτό να είναι κοινό καθήκον και περί αυτού πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να κινηθεί παράλληλα σε δύο πορείε. Από τη μία πλευρά θα συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα. Θα εξετάσουμε τη μεθοδολογία, θα εξετάσουμε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται με πεπισμένη ότι τα κριτήρια είναι αρκετά ακριβή και τα χρησιμοποιούμε πλήρω. Ήταν πολύ αντικειμενική αξιολόγηση βασισμένη σε γνωστά κριτήρια αλλά θα το επεξεργαστούμε το θέμα με τους ενδιαφερομένους κύκλους και η δεύτερη πορεία που θα ακολουθήσουμε, η παράλληλη, θα είναι με τις καταχωρημένες χώρες, εκείνες που θέλουν να εξαλείψουν τον κίνδυνο από την πλευρά τους. Το συζήτησα αυτό με αρκετέ χώρε του καταλόγου που δεν θέλουν να είναι στον κατάλογο. Αυτή είναι μια πρόσκληση που του απευθύνω. Α εργαστούμε ούτω ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνο από την πλευρά σα. Θα πρέπει οι εταίροι μας να μην έχουν πλέον ελλείψεις και κενά. Και πιστεύω ότι είμαστε σαφέστατοι. Αυτή θα είναι μία πορεία που θα ακολουθήσουμε με τις καταχωρημένες ε, χώρες και η άλλη πορεία και άλλη προσπάθεια θα είναι η συνεργασία ε, όσον αφορά την αξιολόγηση των χωρών που είναι στην ομάδα 2 όπου πραγματικά έχουμε τη Ρωσία και άλλες χώρες που αναφέρατε στη συζήτηση. Το μήνυμά μου είναι απευθυνόμενοι προς τα κράτη-μέλη ότι δεν παρετούμε. Ο κινητήρας λειτουργεί, συνεχίζουμε την επεξεργασία διαφόρων θεμάτων, να συμμορφωθούμε με τις ε, υποχρεώσεις που από την νομοθεσία, κάνουμε τα αναγκαία και θα επιστρέψουμε με ένα νέο κατάλογο αργότερα, φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ε, το λόγο έχει εξ ονόματος του Συμβουλίου η κυρία Τσιότ. You heard a lot of criticism from all. Ακούσατε πολύ κριτική από όλες τις πολιτικές ομάδες, πολλές ερωτήσεις. Θέλουμε πραγματικά με ανυπομονησία να ακούσουμε τις απαντήσεις που θα δώσετε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, Παρακολούθησα τις παρεμβάσεις σας ε, και τις παρεμβάσεις της Επιτρόπου. Και θέλω να δράξω αυτή την ευκαιρία για να επανεπιβεβαιώσω τη σημασία στην οποία δίνει η Προεδρία στον ε, αγώνα κατά της ε, χρηματοδότησης της δημοκρατίας και του ξεπλήματος χρήματος. Όπως είπα, το Συμβούλιο θεώρησε ότι υπήρξαν διαδικαστικά προβλήματα, προβλήματα σε σχέση με τη διαδικασία που ακολούθησε η Κομισιόν. Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι η κυρία Γιούροβα είπε ότι ε, πολλοί ε, εξέφρασαν ανησυχίε όσον αφορά τον λίγο χρόνο που αφιερώθηκε στις διαβουλεύσεις καθώς και τη δέσμευσή της ότι η διαδικασία θα βελτιωθεί στο μέλλον. Εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν στον τομέα αυτό. Το Συμβούλιο δεν έχει συγκεκριμένη θέση για την συμπερίληψη συγκεκριμένη χώρα στη λίστα ή όχι. Οι λόγοι για τους οποίους το Συμβούλιο απέρριψε τη λίστα είναι γνωστοί και ήταν, είναι αυτοί που σας παρουσίασα στην αρχική μου παρέμβαση. Αφορούσαν τη μεθοδολογία που ακολούθησε η Κομισιόν, κάτι που ξεκαθαρίζεται και στη δήλωση του Συμβουλίου. Η Προεδρία θα είναι στη διάθεσή σας για να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις για το θέμα αυτό, όπως κριθεί αναγκαίο. Σας ευχαριστώ έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κοέλιο με θέμα σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Κοέλιο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι το Σέγγεν και η ελευθερία διακίνηση είναι μια μεγάλη επιτυχία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μία από τι καλύτερε για του Ευρωπαίου πολίτε και απαιτεί μέτρα τα οποία διασφαλίζουν βέβαια την προστασία των κοινών μα συνόρων, τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών. Απαιτεί όμω επίση και μια πολιτική θεωρήσεων Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που μας επιτρέπει να ελέγχουμε ποιοι μπαίνουν στην επικρατειά μας για να σπουδάσουν, να εργαστούν κτλ. Οπότε το σύστημα θεωρήσεων είναι ένα πολύ βασικό σύστημα και σήμερα περιορίζεται στους ε, τουρίστες. Πρόκειται για θεωρήσεις μικρής ε, διάρκειας. 17 εκατομμύρια θεωρήσεις δόθηκαν το 2017 και όπως είναι προφανές δεν είναι μόνο τουρίστες που μπαίνουν στο Σέγγεν, μπαίνουν και ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι. Άλλοι για επανένωση με τις οικογένειές τους, άλλοι είναι φοιτητέ. Οπότε όλοι αυτοί δεν βρίσκονται σε κανένα ευρωπαϊκό μητρό. Πρέπει να αποφασίσουμε τι ελέγχους θα κάνουμε. Και έπειτα υπάρχει και μια τελευταία κατηγορία που είναι οι μεγάλοι επενδυτές. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια κράτη-μέλη είναι εκτός ΒΙΣ, δηλαδή συστήματος ε, θεωρήσεων μέσα στα πλαίσια του ΣΕΝΚΙΝ. Θα θέλαμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα, το ΒΙΣ. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, θεωρήσεις που εγγράφονται στο ΒΙΣ. Και Γι' αυτό οι σοσιαλιστές άλλαξαν τη θέση τους τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, ε, είπαμε ότι θα πρέπει να εντάξουμε το όλο ζήτημα στο γενικότερο ε, σύστημα θεωρήσεων. Το ίδιο κάνανε μετά και η πράσινη και η γκουε. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι όσοι παραμένουν στο ευρωπαϊκό έδαφος κάτω από 90 ημέρες θα πρέπει να έχουν καθαρά ε, τουριστική βίζα. Κατά, τη... κατά τα άλλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να εγγυηθούμε το καθεστώς ε, θεωρήσεων μέσα στα πλαίσια των αρχών ασφάλειας. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα και γι' αυτό ε, δεν θα πρέπει να χορηγούμε σε έναν Ρώσο, για παράδειγμα, επιχειρηματία χρυσή βίζα για να ζήσει στη Ρουμανία και να εγκατασταθεί. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα επιμέρους ζητήματα και μέσα στα πλαίσια των χρυσών θεωρήσεων. Γι' αυτό η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, βιομετρικά στοιχεία από τα έξι χρόνια και μετά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνεται ε, διακίνηση τουλάχιστον 15.000 ε, μικρών παιδιών στην Ευρώπη ετησίως. Γι' αυτό με το ενισχυμένο ΒΙΣ δεν θα προωθήσουμε θεωρήσεις τύπου shopping Επίσης θα προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας και θα κάνουμε ένα βήμα στα πλαίσια της δικαιοσύνης και της ασφάλειας για να έχουμε μια πραγματική Ευρώπη των πολιτών. Σε Επιτροπής στο λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή τον κύριο Κοέλιο και στους σκιώδεις εισηγητές ε, για το έργο του στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την πρόταση την οποία συζητούμε σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια μη Ευρωπαίοι υπήκοοι εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θεώρηση είτε για ε, μικρό χρονικό διάστημα είτε για μεγαλύτερο. Οι περισσότεροι από αυτούς ε, είναι νόμιμοι ταξιδιώτες που πληρούν τις ε, προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής. Το παρόν σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων μας επιτρέπει να ελέγχουμε στα εξωτερικά σύνορα και στα προξενία ανά τον κόσμο ότι αυτές οι προϋποθέσεις πληρώνται. Βεβαίως, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να καλύψουμε. Με το νέο σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων θα πάψουμε να έχουμε αυτά τα κενά στο σύστημα. Οι αρχέ θεωρήσεων, η συνοριοφυλακή θα έχει τι πληροφορίε που χρειάζονται, θα έχουν τι πληροφορίε που χρειάζονται για να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε εγκληματίε και σε ενδεχόμενου τρομοκράτε να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να εντοπιστούν. Η Ευρώπη, το έχω πει επανειλημμένα, δεν είναι οχυρό και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει οχυρό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος περνάει από τα σύνορά μας. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η Κομισιόν καλωσορίζει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στους στόχους κλειδιά της πρότασής μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στις πιο σημαντικά από αυτά. Πρώτα απ' όλα, η διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών θεωρήσεων στο σύστημα εισόδου-εξόδου, το αιτίας, το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και το ΕΚΛΙΣ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να εντοπίσουμε τη χρήση πολλαπλών ταυτοτήτων και να εντοπίσουμε οποιονδήποτε τελικά αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Επίσης θα κλείσει το κενό πληροφόρηση που υπάρχει για τις ε, άδειες παραμονής και τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας, πληροφορίες ε, τις οποίες δεν μοιραζόμαστε τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέπει τους ε, συνοριοφύλακε και στι αρχέ μετανάστευσης να καθορίσουν γρήγορα κατά πόσο τα έγγραφα που τους ε, παρουσιάζονται είναι ε, έγκυρα και κατά πόσο τα έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι που δικαιούνται να τα έχουν. Θα δείξουν αυτή τη δυνατότητα στι εθνικέ αρχέ επίση να, να μην νομιμοποιήσουν την παρουσία υπηκών τρίτων χωρών που δεν πληρούν τι βασικέ προποθέσει ασφάλεια για την είσοδο και τη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άτομα, παραδείγματο χάρη, που συνδέονται με γνωστές, γνωστά τρομοκρατικά δίκτυα ή γνωστά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό θα κλείσει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε σε, σε επίπεδο ασφάλειας. Τέλος, η συμπερίληψη αντίγραφων των ταξιδιωτικών εγγράφων των ετούντων ε, θεωρήσεων ε, σε αυτή τη βάση δεδομένων. Αυτό το μέτρο από κοινού με την άδεια έτσι ώστε η υπηρεσία συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής να έχουν πρόσβαση στο ΒΙΣ θα διευκολύνει την ταυτοποίηση και την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών χωρίς έγγραφα και αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τρίτες χώρες που ε, δεν ζητούν την επιστροφή τους. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να καταστήλουμε και να προλάβουμε το έγκλημα οι αρχέ επιβολή του νόμου Europol θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων για λόγου πρόληψη, εντοπισμού ή και έρευνα τρομοκρατικών αδικημάτων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Η πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων θα είναι προσβάσιμη και στι αρχέ επιβολή του νόμου για το σκοπό τη έρευνα ή του εντοπισμού ε, ανθρώπων που αγνοούνται ή που έχουν απαχθεί ή που είναι θύματα σωματεμπορίας. Όλα αυτά βέβαια πάντα σεβόμενοι τις αρχές προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί μέρος του πακέτου έξυπνων συνόρων αλλά και της διαλειτουργικότητας. Γι' αυτόν τον λόγο το σκεπτικό και η βάση αυτής της πρότασης θα πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες αλλαγές που προτείνονται στην έκθεση. Πρώτα απ' όλα θυμίζω ότι η συμπερίληψη πληροφοριών για τις άδειες παραμονής στο ΒΙΣ συνδέεται και με το ζήτημα των χρυσών θεωρήσεων. Καταγράφοντας όλα, όλες τις άδειες παραμονής σε ένα σύστημα πληροφοριών, δεν πρόκειται να λύσει βέβαια τις καταχρήσεις σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αυτών των αδειών, όμως προσδίδει μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ των κρατομελών. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το Κοινοβούλιο θέλει να πάει ακόμα παραπέρα αυτό το μέτρο και να δώσει τη δυνατότητα αποθήκευσης και επαλήθευσης στο σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων αυτών των εγγράφων από τη στιγμή της αίτηση για να εξασφαλίσουμε καλύτερο έλεγχο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης ε, του, του εγγράφου της άδειας. Εμείς βλέπουμε θετικά αυτή την πρόταση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τώρα τις, ε, τα πολλαπλά αιτήματα ασφάλειας και ε, παράνομης μετανάστευσης. Δεν πρέπει να ανερώσουμε ε, κάποιες, το σύστημα αυτό αποκλείοντας κάποιες βάσεις δεδομένων από την αναζήτηση. Μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι το έκρης και τα ταξιδιωτικά έγγραφα ε, θα μπορούν να αναφέρονται στο αιτίας και θα ισχύουν πλέον και για το ΒΙΣ αυτά. Είναι ζήτημα συνέπειας και συνέχειας. Οι προδιαγραφές επαλήθευσης των υπηκών τρίτων χωρών που μπορεί να εισέλθουν στην, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όπου δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρηση, δεν πρέπει να είναι πιο αυστηρές από αυτού που δεν έχουν αυτή την υποχρέωση. Τέλο, η Κομισιόν προτείνει να επικαιροποιήσει του κανόνε πρόσβαση στο ΒΙΣ αυτή τη στιγμή. Όμως είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση αυτή θα είναι ισορροπημένη και δεν θα είναι επιζήμια για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Παραδείγματος χάρη, το να προσθέσουμε την υποχρέωση διαβούλευσης των, των βάσεων δεδομένων του ΠΡΙΜ πρώτα, ε, θα είναι, δυσκολεύσει τη διαδικασία. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τη δακτυλοσκόπηση των παιδιών. έχουμε προτείνει να μειωθεί η ηλικία, διότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την εμπορία παιδιών πιο αποτελεσματικά. Είμαι βέβαιος ότι όλοι συμμεριζόμαστε αυτόν τον στόχο. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Και εμείς ανησυχούμε. Η εμπορία παιδιών, το λαθρεμπόριο παιδιών, οι απαγωγές αποτελούν Όμω παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιών δικαιωμάτων. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ετησίω 1.500 ε, με 2.000 ε, παιδιά από τρίτε χώρες που είναι κάτω των 12 ετών είναι θύματα ε, εμπορία και διακίνησης στο χώρο Σέγγεν και 2.500 έω 3.500 για τις ηλικίε 12 έως 15. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά προέρχονται από χώρες που έχουν υποχρέωση Ε, Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και κατεβάζοντα το όριο ηλικία για τα κλωσκόπηση μα δίνει, μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλω να κλείσω τώρα με το πιο σημαντικό σημείο για του πολίτε μα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπω πάντα, θα είναι στην καρδιά όλων των πολιτικών μας και σε ό,τι αφορά τα συστήματα πληροφοριών μας και το σχεδιασμό τους. Όλες οι εκθέσεις για την απόδοση του ΒΙΣ δείχνουν ότι η εφαρμογή του δεν οδήγησε ποτέ σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ανησυχίες περί δεδομένων. Ούτε μία προσφυγή δεν υπήρξε κατά το Συστήμα πληροφοριών θεωρήσεων μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας. Και πήγαμε ένα βήμα παραπέρα σε ό,τι αφορά δηλαδή την προστασία δεδομένων εξ αρχής. Βεβαίω, κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τι προδιαγραφέ αυτέ, παραμένοντα όμω αποτελεσματικοί, χωρί δηλαδή να αποκλίνουμε από του βασικού μα στόχου. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και αναμένω με ανυπομονησία τη συζήτησή μα. Επίτροπε, το λόγο εκ μέρου τη Επιτροπή Προπολογισμού έχει ο κύριο Κέλμελ για ένα λεπτό.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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Η Επιτροπή των Προϋπολογισμών ε, στηρίζει πλήρως αυτά που είπε ε, ο εισηγητής. Σήμερα τον υπάρχουν συμβατά συστήματα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Κυρίως ε, στο θέμα της διέλευσης συνόρων και στο θέμα των θεωρήσεων πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι απάτες σε θέματα ταυτότητας. Αλλά πρέπει επίσης να μπορούμε να εντοπίζουμε με μεγαλύτερη ευκολία τις ε, ταυτότητες. Αυτό αφορά βεβαίως και τον αγώνα κατά της ε, τρομοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν επενδύσεις. Με βάση τους υπολογισμούς μας ε, χρειάζονται 461 εκατομμύρια σε 9 χρόνια. Υψηλό το ποσό, αλλά είμαι πεπισμένος ότι και εμείς και οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά τα χρήματα θα έχουμε καλύτερη ασφάλεια. Άρα δηλαδή θα είναι καλά επενδεδημένα κονδύλια. Πρέπει να είναι σαφές ότι μόνο για το 19 και το 20 υπάρχουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού στο νέο πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει όμως να προβλεφτούν εκ νέου αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κάνω έκκληση να γνωρίζει το Κοινοβούλιο ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτό το πρόγραμμα πρέπει τα κονδύλια να υπάρχουν και στον επόμενο προπολογισμό. Γιατί αλλιώ αλλιώς ε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει ο κύριο Ράντεφ για 1,5 λεπτό. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ε, το σύστημα των θεωρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εντοπίσουν κατά πόσον οι θεωρήσεις ισχύουν και είναι και γνήσιες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τις ε, βραχυπρόθεσμες θεωρήσεις που έχουν ε, νομοθετηθεί και αυτό είναι ένα κενό. Ε, χαιρετίζω τις προτάσεις. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και μακροπρόθεσμες θεωρήσεις. Αυτά λοιπόν τα έγγραφα αποτελούν επίσης μία δυνατότητα για την ελεύθερη μετακίνηση στο χώρο του Σέγκεν. Ε, χρειαζόμαστε και τις μακροχρόνιες θεωρήσεις για να αντιμετωπίσουμε και την παράτυπη ε, μετανάστευση. Πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο θεωρήσεις ισχύουν και είναι και γνήσιες. Η αναθεώρηση του συστήματος ΒΙΣ είναι απαραίτητη, σημαντική η διαλειτουργικότητα και η εναρμόνιση ε, τα συστήματα ασφαλείας ε, τα οποία ε, προσφέρουν πληροφορίες θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό χωρίς βεβαίως να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και των δεδομένων τους. Τέλος, ε, θα ήθελα να καλέσω ε, το Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων να λάβει μια θετική απάντηση όσον αφορά την ε, συμπερίληψη της Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το σύστημα των θεωρήσεων και να συμβάλλουμε σαν διαφυλάστε η ασφάλεια στην Ευρώπη. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Νίντερ Μίλλερ. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο, για την ε, επικοδομητική του εργασία, αναζήτησε συμβιβασμού, βασίστηκε στη συνεργασία. Πιστεύω ότι το σύστημα των θεωρήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πολιτική, στην ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, να ε, προχωρήσουμε σε αυτό το σύστημα γιατί κάθε χρόνο εκδίδουμε εκατομμύρια θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση που προτείνεται έχει ως κύριο στόχο να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών στα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί ε, όσον αφορά τις προκλήσεις ασφάλειας πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να λειτουργούν τα συστήματα αποτελεσματικότερα. Και σε τελική ανάλυση τα συστήματα ε, πρέπει να ενισχύουν την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμίσης η δική μου πολιτική ομάδα θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ε, η άποψη του αρμοδίου για την προστασία δεδομένων, κυρίως όσον αφορά τις μακροχρόνιες θεωρήσεις. Και οι δύο εκθέσεις υπογραμμίζουν ε, την αναγκαιότητα, την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Η προτινόμενη ε, νομοθεσία σχετίζεται με το ότι τα συστήματα πρέπει να είναι συμβατά, γιατί κάθε σύστημα ε, μπορεί να επηρεάσει συστήματα άλλων τρίτων χωρών. Έχουμε λοιπόν θέσει επανειλημμένα το θέμα της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Συνεχίζουμε να το πράττουμε. Ε, αυτό βέβαια ε, σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Νομίζω ότι επιτύχαμε μια ικανοποιητική συμβαστική λύση. Η πρόταση δεν παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, βελτιώνει την ασφάλεια, την ενισχύει και έτσι επιτυχάνει το στόχος. Στον το λόγο έχει η κυρία Στίβενς για ένα λεπτό. Voorzitter, collega's. Κύριοι συνάδελφοι, το σύστημα ΒΙΣ, το σύστημα ε, πληροφοριών για τις θεωρήσεις, θέλει να καταπολεμήσει την ε, παράνομη μετανάστευση και έτσι θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών για τη διέλευση των εξωτερικών μας σύνορων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε 60 εκατομμύρια θεωρήσεις που χορηγούνται κάθε χρόνο για βραχυχρόνια διαμονή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται αυτόματη διασταύρωση στοιχείων με άλλα συστήματα πληροφοριών καθώς ε, και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικό αυτό το σύστημα. Το κείμενο που έχουμε ενώπιον μας είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για την επόμενη θητεία. και Δημοκρατών, το λόγο έχει κύριος για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 48 εκατομμύρια ε, είναι τα αιτήματα θεωρήσεων και 140 εκατομμύρια οι δακτυλοσκοπήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε ένα αποδοτικό σύστημα. Με βάση την έκθεση Κάρλος Κοέλιο, τον οποίο θα ήθελα να συγχαρώ για την εργασία του, το σύστημα θα είναι ακόμα πιο αποδοτικό. Θεωρούμε ε, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και της άδεια διαμονής ε, καθώς και τις μακροχρόνιες θεωρήσεις διότι δεν γίνονται ανταλλαγές πληροφοριών για αυτές τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να καλύψουμε ολόκληρο το χώρο Σέγγεν και να υπάρχει διαφάνεια ως προς την πώληση θα μπορούσα να πω των θεωρήσεων αυτών καθώς και των μακροχρόνιων των αδειών μακροχρόνιας διαμονής. Επίσης θα πρέπει να εγγραφούν τα στοιχεία της Europol στο ΒΙΣ. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουμε και τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να είμαστε σίγουροι ότι προβλέπεται επιστροφή. Θα πρέπει επίσης να γίνεται η δακτυλοσκόπηση από τα 6 χρόνια ηλικία σε σχέση με τα 12 που ίσχυαν μέχρι τώρα για να υπάρχει καλύτερη προστασία των ανηλίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, το 40% των παιδιών που αποτελούν ε, αντικείμενο διακίνησης είναι κάτω των 12 ε, ετών. Επίσης, θα πρέπει οι αιτήσει θεωρήσεων να βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία ως προς τους εμπλεκόμενους κινδύνους για να μην υπάρχει και άρνηση χορήγησης εκεί που δεν χρειάζεται. Ε, κάθε επιτυχία σου εύχομαι Κάρλος και θα σας υποστηρίξουμε. Εκεί αριστερά στο λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Βερζιά. Θα είμαι λίγο μόνη τώρα εδώ. Φαντάζομαι το 2004 δημιουργήθηκε, το 2014 τέθηκε σε ισχύ. Το ΒΙΣ, λοιπόν, όπως και ο κώδικας ε, θεωρήσεων, είχε ω στόχο να διευκολύνει τι θεωρήσεις. Από το 2014 όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ λυπηρά. Μιλάμε πλέον για γενικευμένο έλεγχο και σταστηματικό φακέλωμα. Ε, συγχαίρω τον εισηγητή μας που μας βοήθησε να αφαιρέσουμε μια φορά από ζητήματα αρκετά προβληματικά, όπως ε, το θέμα της Interpol, όπου κάποιες, κάποιες χώρες μπορούν έτσι να πιάσουν ε, αντιφρονούντες που έχουν, που έχουν διαφύγει, όπως με τη Σαουδική Αραβία πρόσφατα. Κάποιοι μπερδεύουν λοιπόν τα υγειονομικά, την, ε, ε, τα μεταναστευτικά, τα τρομοκρατικά. Δεν είμαστε υπέρ ε, της, ε, των να ασχολούμαστε με τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας. Η επικουρικότητα λοιπόν έχει πάει περίπατο και δεν συμφωνούμε στο να πέσει η, ηλικία από το, για την δεσλογοσκόπηση των παιδιών από τα 16 στα 12. Πάει και η αναλογικότητα έτσι. Δεν είμαστε υπέρ της ασφάλειας πάση θυσία με αυτό το τεράστιο κόστος. Για, για, για αυτά τα θέματα βέβαια πάντα υπάρχουν χρήματα ο κατάλογος των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για ένα λεπτό. Señor presidente, comisario debatimos aquí en el pleno del Parlamento. Κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, συζητήσαμε εδώ το νέο σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων. Περί τίνο πρόκειται να επιτρέψουμε τη διασύνδεση των συνοριοφυλάκων των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ένωσης με τα προξενία των κρατών μελών σε όλο τον κόσμο έτσι ώστε να μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να δίνουμε πληροφορίες για όσους ετούνται θεώρηση έγκεν όταν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια μέσω βιομετρικών ε, συγκρίσεων, βιομετρικών στοιχείων, δακτυλοσκοπικών ε, ευρημάτων. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα επιτρέπει τη διασύνδεση μέσω των νέων τεχνολογιών και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων που σχετίζονται με τους ετούντες άσυλο και τους ετούντες θεώρηση μάλλον ε, και τις απειλές για την ασφάλεια των κρατών μελών. Από την σοσιαλιστική ομάδα εμείς έχουμε συνεισφέρει με εγγυήσει σε ό,τι αφορά την αρχή της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και εγγυήσει βέβαια σεβασμού των δικαιωμάτων των θεμελιών δικαιωμάτων και του σχετικού χάρτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων. Ε, το σημαντικό όμως είναι να μην προχωρούμε μόνο σε επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε ένα συνολικό σύστημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, thank you. Uh, Commissioner, colleagues, uh, I welcome the θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω το σύστημα αυτό για τις θεωρήσεις καθώς και τις ε, μακροχρόνιες θεωρήσεις. Ως ε, μέλος των σοσιαλιστών με απασχολεί το θέμα της ιδιωτικότητας σε σχέση με την εξέταση των θεωρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα, αλλά αυτό θα οδηγούσε σε παράνομες ε, ε, μεταφορές στοιχείων. Βεβαίως μπορούμε να αποτιμήσουμε κινδύνους, αλλά εκθέτουμε ευαίσθητα στοιχεία σε μεγάλους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνδεσιμότητα με άλλα συστήματα. Καμία ε, επιχείρηση, για παράδειγμα, δεν μπορεί να προωθήσει τη συνδεσιμότητα αυτών των στοιχείων. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα ε, ζητήσουμε από μία ειδική επιχείρηση να ασχοληθεί με τη συνδεσιμότητα. Δικασία του Κατσιδιάη, έχω δεχθεί δύο αιτήματα, γίνονται και τα δύο αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις πραγματικά χρειάζεται αρκετές βελτιώσεις και νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτή την κατεύθυνση πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. όμως κύριε Αβραμόπουλε επιτρέψτε μου να σας θέσω ένα θέμα γιατί φοβάμαι ότι σε λίγο όσοι ερχόμαστε με αεροπορικές πτήσεις από την ελλάδα στο βέλγιο θα χρειαζόμαστε βίζα. σας είχα καταγγείλει το απαράδεκτο φαινόμενο της καραντίνας που είχαν επιβάλει στα γερμανικά αεροδρόμια αλλά και στο αεροδρόμιο των βρυξελών και είχα λάβει απάντηση στο θέμα αυτό από εσάς στις 23 Νοεμβρίου ότι το είχατε βρει ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Σας λέω λοιπόν ότι στις 19 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου ξαναεπαναλήφθηκε αυτό το σύστημα καραντίνας και εκεί στη μια περίπτωση εμφανίστηκαν δίθεν αστυνομικοί στην άλλη περίπτωση εμφανίστηκαν δίθεν τελωνιακοί και εγώ αλλά και ο κύριος παπαδημούλης που ήμασταν στην ίδια πτήση και άλλοι ευρωβουλευτές είχαμε την δυσμενή τύχη ατυχία αν θέλετε να υποβληθούμε σε διαβατηριακό έλεγχο. είναι νόμιμο αυτό; μπορεί να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία στο αεροδρόμιο των βρυξελών; θέλουμε μια απάντηση κύριε επίτροπε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. σε λίγο θα χρειαζόμαστε βίζα από την ελλάδα για τις βρυξέλλες. ευχαριστώ. Ε,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 Πρόκειται για ένα σύστημα πάρα πολύ επίμαχο, πάρα πολύ δαπανηρό, ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται θα χρησιμοποιείται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες ανάγκες. Ε, οι θεωρήσεις ε, θα μπορούσαν να είναι σε διαφορετικές ε, περιπτώσεις για διαφορετικά άτομα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία. Η Τρομοκρατία όμως ε, προκύπτει κυρίως από Ευρωπαίους, αν θέλετε, πολίτες δεύτερης, τρίτης ε, γενιάς και μετά υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχουμε αυτούς που έρχονται σε εμά. Ναι, αλλά εκατομμύρια έχουν έρθει εδώ, πολλούς μάλιστα τους καλέσαμε να έρθουν και αυτοί είναι ήδη εδώ. Φαίνεται κατά την άποψή μου ότι πρόκειται για ένα πείραμα πάρα πολύ ε, δαπανηρό το οποίο δεν θα οδηγήσει πουθενά. Το λόγο έχει εκ μέρους της Επιτροπής, κύριε Σαβραμού. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω το γεγονός ότι μέσα σε ένα μόνο χρόνο ε, κατορθώσαμε ε, ή κατορθώσατε εσείς ε, να επιτύχετε τη συμφωνία με το Συμβούλιο για το Ιουλίζιο, το SSS, το ΕΤΙΑΣ και τις διατάξεις περί συμβατότητας. Τα συστήματα θεωρήσεων μαζί με το σύστημα ΕΤΙΑΣ και μαζί με άλλα συστήματα από κοινού με μια νέα πλατφόρμα για τρίτους, για τρίτους, τρίτων κρατών που επισκέπτονται την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύστημα θα κλείσει το κενό που υπάρχει, ε, κενά ασφαλείας ε, αυτό αφορά τόσο τους επισκέπτες μικρής όσο και μακράς διάρκειας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό τα συστήματα να συγχρονιστούν στον βαθμό του δυνατού. Και είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι το σύστημα θεωρήσεων θα πρέπει να συμφωνήσει